2014 και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους. Το ΕΛΚ, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι μου ζήτησαν ε, να ε, διορίσουν άτομα και να αλλάξει η σύνθεση κάποιων επιτροπών και αντιπροσωπιών. Η λίστα είναι στην διάθεσή σας. Εάν μέχρι το τέλος συνεδρίας δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, εγκρίνονται αυτές οι αλλαγές. Επίσης